που προασπίζει τις ε, θεμελιώδεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και απέναντι στο Αφγανιστάν. Ευχαριστώ κύριε Αλμούνια. Έχω δεχτεί πέντε προτάσεις ε, ψηφίσματος ε, των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Ε, ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει στη συνέχεια. Τώρα ακολουθεί η συζήτηση για την κατάσταση των γυναικών στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν. Θα δώσω το λόγο στου συντάκτε. Πρώτο ο κύριο Τάνοκ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κατάσταση των γυναικών στο Πακιστάν και Αφγανιστάν παραμένει σοβαρή. Παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά των γυναικών δυστυχώ είναι ψωμοτήρι και πολύ συχνά οι αρχές τις ανέχονται θα πρέπει ιδιαίτερα στο Πακιστάν να ληφθεί υπόψη αυτό και το ε, κυβέρνηση να ε, μην ε, επιτρέπει την ατιμορρησία. Επίσης και οι ακροτηριασμοί θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο Αφγανιστάν. Έχουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη περίπτωση και θνησιμότητα των μητέρων στον κόσμο. Επίσης στο Αφγανιστάν επιτρέπεται σε κάποιες περιοχές η εκτέλεση εγγύων. Θα πρέπει να σταματήσει αυτό. Βεβαίω είναι κατά ε, της ε, Χάρτας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του ΟΗΕ. Παρά την οικονομική και τεχνική ενίσχυση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν, οι γυναίκες δυσκολεύονται να φτάσουν στη στοιχειώδη εκπαίδευση. Υπάρχει πολύ βαθιά διάξηση βάρους των γυναικών δεν γίνονται προσπάθειες ε, για την ισότητα ούτε πρόσληψη ε, σε θέσεις επιρροής όπως είναι η δικαιοσύνη ή η Βουλή. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση ε, βιώσιμη πριν αποσυρθούν το 2014 τελικά οι δυνάμεις της ΆΙΣΑΦ και του ΝΑΤΟ. Εμείς πιστεύουμε ότι εκτός από τα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι χώρες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να βοηθάει με προγράμματα που προωθούν τα δικαιώματα των γυναικών στις δύο αυτές χώρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκένγκερ Ντεόντεμπεργκ για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Φαίνεται απίστευτο που στον 21ο αιώνα υπάρχουν ακόμη χώρες που ουσιαστικά απαγορεύουν στις γυναίκες να συμμετέχουν ε, ενεργώς στον δημόσιο βίο, πολιτικό και κοινωνικό. Στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν οι γυναίκες δεν έχουν καμία δυνατότητα να εξελιχθούν, να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητές τους και πολλές φορές είναι θύματα κυρώσεων, ποινών, ε, διώξεων. Ε, διώκονται καθημερινά οι γυναίκες στις χώρες αυτές. Λόγω λοιπόν του καθεστώτος, μετά το καθεστώτος των Ταλιμπάν, η κατάσταση του Αφγανιστάν έχει βελτιωθεί ελαφρώς. Όμως το Πακιστάν έχει αντιθέτως επιδεινωθεί. Λόγω των μέτρων που προβλέπουν διακριτική μεταχείριση, Οπότε, προφανώ, χρειάζεται αναθεώρηση των δικαιωμάτων προστασία των γυναικών σε χώρε όπω αυτέ θα πρέπει πρώτα απ' όλα να διασφαλίζεται ο έντιμο βίο και η αξιοπρέπειά του, η προσωπική του εξέλιξη και η επαγγελματική του εξέλιξη, η ασφάλεια στα σχολεία και στο χώρο εργασία. Θα πρέπει να προσφέρει υποστήριξη η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτέ τι χώρε. Όχι μόνο να εκφράζουμε το θυμό μα, αλλά να καλούμε για την ίση μεταχείριση των δύο φύλων. Ευχαριστώ κύριε Γκέρνγκερ. Ο κύριος Ρωμέβα Ιρουέντα για δύο λεπτά παρακαλώ. Δέκα χρόνια μετά τη λεγόμενη διάσκεψη του Πέτερσμπεργκ για το Αφγανιστάν το 2001 που έθεσε τα θεμέλια της συνεργασίας διεθνούς κοινότητας με το Αφγανιστάν είναι γεγονός ότι έχει γίνει κάποια πρόοδος για τις γυναίκες. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, πάνω από 4 εκατομμύρια κορίτσια πηγαίνουν στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο, 70% ε, και 25% ε, το μελών του Κοινοβουλίου είναι γυναίκες και 70% υποτίθεται ε, στη δίκηση. Αλλά παραμένει πολύ μεγάλη η μετρική θνησιμότητα και ο αναλφαβητισμός. Ε, αναγκαστική γάμη μεταξύ αυτών και για παιδιά, διακίνηση, σώματεμπορία, Ε, πολλές φορές ε, δίνεται ή πωλείται ένα κορίτσι, μια γυναίκα προς επανόρθωση εγκλήματος ως ποινή. Και είναι πολύ συχνό φαινόμενο οι Ταλιμπάν να τιμωρούν τις γυναίκες. Οι Αφγανές γυναίκες γνωρίζουν όλο και περισσότερες επιθέσεις. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό ζητούμε ε, τις αρχές ασφαλείας να τις εκπαιδεύουμε όχι μόνο για την αντιμετώπιση των εξεγερθέντων αλλά για να επιβάλλουν τον νόμο και την τάξη. Και ας θυμηθούμε ότι οι γυναίκες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην κοινωνία και να είναι ηγέτες των προγραμμάτων και να συμμετέχουν στην εκπόνηση αυτών. Για το Πακιστάν, αντίστοιχη κατάσταση και θα πρέπει να την καταγγείλουμε. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι σε ορισμένες περιφέρειες οι αρχές δρούν με πολύ ε, αντίστοιχο τρόπο με κίνηση του Αφγανιστάν. Γι' αυτό ζητούμε από την κυβέρνηση του Πακιστάν να επαναφέρει τα όσα ίσχυαν το 1973 για την ισότητα μετά το πραξικόπημα του 1977 ε, και να μην υπάρχουν διακρίσεις με βάση το φύλλο. Ευχαριστώ κύριε Ρωμέβα Ιρουέντα. Για ένα λεπτό ο κύριος Μέρφη. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ και δέκα χρόνια το, η προστασία των γυναικών ε, χρησιμοποιήθηκε ω πρόσχημα για τον πόλεμο κατά του Αφγανιστάν. Όμω η κατάσταση των γυναικών παραμένει πάρα πολύ άσχημα. Έχουν το χαμηλότερο επίπεδο αλφαβητισμού στον κόσμο, 13% και μόνο 5% μπορούν να πάνε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Χειρότερο από ότι, καλύτερα μάλλον από ότι ήταν το, υπό το καθεστώ των Καραλμπάν, αλλά πολύ χειρότερα από ότι το 2005. Ε, μεταξύ του 60 και του 80% των γάμων είναι, είναι καταναγκαστικοί και υπάρχουν ε, πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά οικιακή βία. Είναι πολύ επικίνδυνο μέρο λοιπόν ε, στον κόσμο αυτό για να είναι κανεί γυναίκα. Οι χώρε αυτέ, το Πακιστάν και το Αφγανιστάν. Το παράδειγμα μια γυναίκα που βιάστηκε όταν ήταν 19, ε, έμεινε έγκυο και καταδικάστηκε, φυλακίστηκε για το έγκλημα τη εξαναγκαστική μοιχεία. Χθε μόλι απελευθερώθηκε ενώ αντιμετώπιζε την απειλή 12 ετούς εδώ υπάρχουν πολλέ τέτοιε γυναίκε που έχουν φυλακιστεί για ανάλογα έγκληματα. Χρησιμοποιείται όμω και ω πρόσχημα η κατάσταση αυτή για να συνεχίζεται η κατοχή τη χώρα. Έχει ανακοινωθεί η απόσυρση των στρατευμάτων ή για αποχώρησή του, όμω θα πρέπει να ε, προωθηθούν όλοι οι υπερασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, κύριο Πρέντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα μιλάμε για χώρες όπως το Πακιστάν και το Αφγανιστάν. Σε χώρες αυτές θα πρέπει να εντοπίσουμε κάποια στοιχεία που θα μπορούσαν να είναι και θετικά. Στο Αφγανιστάν, λόγου χάρη, κάποιες γυναίκες έχουν διοριστεί σε θέσεις ευθύνη. Πρόσφατα, η Κουνάζ όμως καταδικάστηκε σε φυλάκιση. Στο Πακιστάν επίσης η έγκριση κανόνων για την μη βίαιη συμπεριφορά των γυναικών Όλα αυτά είναι ενθαρρυντικά σημάδια. Όμω και στι δύο χώρε παραμένουν σοβαρά, σοβαρές ανησυχίες. Στο Αφγανιστάν, η συζυγική βία, όπως και στο Πακιστάν, παραμένουν. Από την άλλη, στο Αφγανιστάν, ο λιθοβολισμός για την παραβίαση κάποιων κοινωνικών κανόνων ισχύει ακόμα, ενώ στο Πακιστάν οι γυναίκε πέφτουν θύματα εγκλημάτων τιμή, όπω λέγονται ή ε, πολλές φορές εξαναγκάζονται να ε, αλλάξουν τη θρησκεία τους. Αυτές είναι πρακτικές τις οποίες πρέπει να τις καταγγείλουμε και εδώ. Ευχαριστώ κύριε Πρέτα. Ένα λεπτό η κυρία Νικολάη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το ψήφισμα αυτό ναι, με να απευθύνεται σε δύο χώρες με διαφορετική κατάσταση σε τεφορά αφορά τις γυναίκες έχει κάποια όμως κοινά σημεία. Πρώτα απ' όλα, αντιμετωπίζουμε δραματική κατάσταση σε ό,τι αφορά την ισότητα, ε, τη δικαιώματα των γυναικών, τη βία κατά των γυναικών. Και μιλώ ιδίως για το Πακιστάν. Σε ό,τι αφορά το Αφγανιστάν, πρέπει να παραδεχθούμε ότι έχει βελτιωθεί ελαφρώς η κατάσταση, οικονομικής τουλάχιστον πλευράς. Ε, το πρόσφατο Αφγανικό Σύνταγμα προβλέπει την ισότητα των, ε, ευκαιριών και υπάρχει και ένας ε, νόμος ε, για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών από το 2009 που πλέον εφαρμόζεται. Επίσης νομίζω ότι και η εκπροσώπηση των γυναικών έχει βελτιωθεί πρόσφατα, αλλά πρέπει να παραδεχθούμε ότι τα πράγματα θα γίνουν πιο δύσκολα όταν αποσυρθούν τα διεθνή στρατεύματα από το Αφγανιστάν γιατί νομίζω ότι ό,τι θετικό ε, δημιουργήθηκε του τελευταίου μήνε και χρόνια κινδυνεύει να χαθεί. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να εντείνει τα προγράμματα συνεργασία για να διατηρηθούν τα πράγματα στη σημερινή κατάσταση. Ευχαριστώ κύριε Νικολάη. Εδώ ήταν οι συντάκτε, Ακολουθούν οι ομιλητέ εξ ονόματο των πολιτικών ομάδων. Ένα λεπτό, ο κύριο Πόσελτ. Κύριε Πρόεδρε, και οι δύο χώρε είναι πολύ διαφορετικέ, παρότι γείτονε αλλά και μεγάλες διαφορές στο εσωτερικό των χωρών. Το Πακιστάν είχε γυναίκα αρχηγό κράτους πολύ πριν ε, ε, τη Γερμανία, μάλλον ε, πρωθυπουργό. Και στο Αφγανιστάν υπάρχουν γυναίκες κυβερνήτες. Υπάρχουν όμως και περιφέρειες όπου κυβερνούν οι φυλές και οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να πάνε ούτε στο σχολείο τα κορίτσια ούτε στο γιατρό καν. Αυτές τις κατάφορες διαφορές μπορούμε να τις ξεπεράσουμε με μεταρρυθμίσεις, όχι με ιδεολογία. Γι' αυτό απέτυχε η προσπάθειά μας στο Αφγανιστάν. Γιατί θέλαμε ε, ε, χιλιετίες να τις ξεπεράσουμε με ένα άλμα. Αυτό δεν γίνεται. Ούτε στην Ευρώπη έγινε. Πού να γίνει στο Χιντοκούς. Γι' αυτό θα πρέπει να συνηθίσουμε ότι οι χώρες αυτές έχουν τη δική τους εξέλιξη και χρειάζεται υπομονή και μόνιμη υποστήριξη και όχι με ε, στρατεύματα ούτε πατάς ένα κουμπί και αλλάζει κοινωνία. Ευχαριστώ κύριε Πόσελτ. Η κυρία Σένισιν για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Σύμφωνα με το Reuters, το Αφγανιστάν είναι πρώτο σε ό,τι αφορά την παρέμβαση των δικαιωμάτων των γυναικών ε, στον κόσμο. Τρίτη χώρα ε, στην κατάταξη είναι το Πακιστάν. Εγκλήματα τιμή, ε, κακοποίηση γυναικών είναι στην ημερήσια διάταξη. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με την προσέγγιση του κράτους, διότι το θρήσκευμα, η θρησκεία που επικρατεί είναι αυτή η οποία ουσιαστικά καταπιέζει τις γυναίκες. Πολύ Πολλές γυναίκες έχουν καταδικαστεί είτε για μοιχεία είτε γιατί έφυγαν από το σύζυγό τους τα λεγόμενα ηθικά εγκλήματα. Πολλές χιλιάδες γυναίκες έχουν ε, ε, υποστεί βιασμούς, ε, σεξουαλική ή, άλλου, ή ψυχολογική πίεση, καταπίεση. Δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση όμως στο Αφγανιστάν, έχει επιδεινωθεί. Οι νόμοι ίσα ίσα αυξάνουν τι επιθέσει των ε, ανδρών κατά των γυναικών και πρέπει να είμαστε κατά. Ευχαριστώ κυρία Σενσίν. Η κυρία Ογιούλαντ για ένα λεπτό παρακαλώ. Δυστυχώ απουσιάζει. Η κυρία Βερζιά για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για άλλη μια φορά εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για την κατάσταση στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν και ιδιαίτερα ως προς τα δικαιώματα των γυναικών. Το έχουμε ξαναπεί. Οι χώρες αυτές είναι θλιβεροί πρωταγωνιστές και πρωταθλητές ε, στα εγκλήματα κατά των γυναικών, δολοφονίες, στα εγκλήματα τιμής. Είναι μακρύς ο κατάλογος. Οι συνάδελφοί μου έδωσαν παραδείγματα. Δεν πιστεύω ότι τα στρατεύματα στο Αφγανιστάν βοήθησαν τις γυναίκες σε κανένα βαθμό. Ούτε ότι η απόσυρσή τους ε, θα επιδεινώσει το παραμικρό. Θα έλεγα όμως ότι μάλιστα θα πρέπει να πιέσουμε τις χώρες αυτές για να αλλάξουν τα πράγματα και όχι μόνο από νομικής πλευράς. Έχουμε συμφωνίες, εταιρικές σχέσεις με τις χώρες αυτές. Ας τις χρησιμοποιήσουμε με το σωστό τρόπο και προς το συμφέρον και όφελος των πολιτών, των αμάχων, υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Ας βγάλουμε τα διδάγματα από τα σφάλματα του παρελθόν μας, ιδιαίτερα στο Μαγκρέμπ. Ας ενεργοποιήσουμε τη ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και τότε θα δρέψουμε καρπούς. Ευχαριστώ κύριε Βερζιά. Ο κύριος Πάσκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η θέση των γυναικών στις Ισλαμικές χώρες είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και επιβαρύνεται και από μακροχρόνιες παραδόσεις, ειδικά σε απομονωμένες περιοχές ή σε περιοχές που κατέχονται από στρατιωτικές θρησκευτικέ ομάδες. Μεσαιωνικές πρακτικές εφαρμόζονται ακόμη θα πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε στον πληθυσμό των χωρών αυτών, να προσπαθούμε να τους ε, στρέψουμε προς έναν εξυγχρονισμένο τρόπο ζωής. Είναι καθήκον της Ένωσης να προστατεύσει τις γυναίκες, οι οποίες είναι θύματα συζυγικής βίας λόγου χάρη, ταπεινώσεων, εξευτελισμών. Η ανθρωπιστική μας βοήθεια πρέπει και αυτό να λάβει υπόψη και να στοχεύσει συγκεκριμένα τις γυναίκες. Θα πρέπει εδώ να υπάρξει διαρκής πίεση κατά των ε, αρχών των χωρών αυτών, ώστε να προσπαθήσουν να περιορίσουν τις πρακτικές κατά των γυναικών. Θα πρέπει οι κρατικές αρχές να είναι προσωποποίηση ενός πολιτισμένου τρόπου ζωής, μιας ευνομούμενης ε, διαβίωσης και να μην διαρκούν οι μακροχρόνιες παραδόσεις που είναι άνθρωπες. Ευχαριστώ κύριε Πάσχα. μισή λεπτό είχατε, αλλά δεν πειράζει. Ευχαριστώ. Αυτοί ήταν οι ομιλητέ εξ ονόματο των ομάδων. Έχουμε άλλους τρεις τώρα, την κυρία Κόρχολα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι ε, βιοπραγίες κατά των γυναικών στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν είναι κάτι που μπορούμε δύσκολα να κατανοήσουμε. Ο νόμος που επικρατεί εκεί είναι κάτι ανάμεσα σε θρησκευτικό και μη θρησκευτικό νόμο με άφρονα τρόπο εφαρμόζεται η σαρία. Σε περίπτωση μοιχείας ε, πταίει πάντα η γυναίκα. Δεν είναι σωστή αυτή η ερμηνεία. Και στις δύο χώρες οι ε, διαφορές είναι μεγάλες. Υπάρχουν πολλές γυναίκες ενεργές στην κοινωνία των πολιτών στις πόλεις, αλλά στην Ήπεθρο οι γυναίκες ζουν μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα. Ας πούμε στις πόλεις υπάρχουν γυναίκες ε, έμποροι. Όχι όμως και στην Ήπεθρο. Μπορεί να βελτιώθηκε η κατάσταση, αλλά δεν ξέρουμε αν θα είναι μόνιμη και η φόρος η κατάσταση, γιατί ε, υπάρχουν κανόνες που ισχύουν ανάλογα με την περιοχή και ανάλογα με την κοινωνική τάξη. Και οι στατιστικές δεν είναι πάντα σωστές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Κρέτσου ευχαριστώ πρόεδρε όπως είπαν οι συνάδελφοι υπήρξαν κάποιες βελτιώσεις στο αφγανιστάν ωστόσο ε, είναι παράλογο που η κατάσταση των γυναικών στο Αφγανιστάν παραμένει σχεδόν η ίδια με το τι γινόταν πριν από μία δεκαετία, όταν υπεγράφει η συμφωνία για τη δημιουργία τη μεταβατική κυβέρνηση υπό την προεδρία του Κατσάι. Εδώ το ποσοστό θνησιμότητα και τη παιδική θνησιμότητα ε, έχουν ε, επιδεινωθεί. Και οι τακτικέ επιθέσει κατά των γυναικών και των κοριτσιών που θέλουν να πάνε στο σχολείο, στο σχολείο ή να συμμετάσχουν στο δημόσιο βίο είναι κάτι το συνεχέ. Εδώ λοιπόν υπάρχει λυπή ε, εκπροσώπηση των γυναικών στο κοινοβούλιο και το δημόσιο βίο και οι Αφγανέ παραμένουν θύματα συζυγική ε, βία, ε, καταναγκαστικών μάλλον γάμων, δικαιο, δικαστικής και αστυνομικής διακριτικής μεταχείρισης. Πρόσφατα επεισόδια έκρηξη με θύματα κορίτσια στο Αφγανιστάν είναι χαρακτηριστικό του τι συμβαίνει με τι γυναίκε στη χώρα αυτή. Η εταιρική μα σχέση βεβαίω θα, παραβε... θα υπονομεύεται από μια τέτοια διαρκή βίαιη υπονόμευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τη χώρα αυτή. Οι αρχέ λοιπόν του Πακιστάν και του Αφγανιστάν πρέπει να λάβουν μέτρα. Ευχαριστώ κύριε Κρέτσο. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αρχές Δεκεμβρίου η διεθνής κοινότητα συναντήθηκε στη διάσκεψη του Μπαντού με τις αφγανικές αρχές. Δεσμεύτηκε το Αφγανιστά να συμπεριλάβει και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο σύνταγμά του, συμπεριλαμβανομένης και της ισότητας ανθρώπων γυναικών, την οποία θα πρέπει να καλωσορίσει και να υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2014 οι συμμαχικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από το Αφγανιστάν και το Αφγανιστάν θα έχει πλήρη ανεξαρτησία να κυβερνάει. Γίνεται ένας διάλογος ε, ειρηνευτικό μεταξύ τη κυβέρνηση και κάποια στοιχεία των Ταλιμπάν, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε επιδείνωση των δικαιωμάτων που κατέκτησαν οι γυναίκε. Και εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να του υποστηρίξουμε. Σα ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι του Ρουντ Χόιστάιν. Αυτοί ήταν μιλητέ που είχαν ζητήσει το λόγο. Ερχόμαστε στη διαδικασία Κατσιά, η κυρία Γκόμε. Πρόεδρε, δεν θα ξεχάσω ποτέ τις γυναίκες που αυτοπερπολήθηκαν και τις οποίες επισκέφτηκα στο Ιράκ το 2008 και τις γυναίκες που βγήκαν από τις φυλακές του Αφγανιστάν αποδρώντας από καταπιεστικές οικογένειες και μια αστυνομία ένα δικοστικό σύστημα που ασκεί δικαιωτική μεταχείριση εναντίον τους. Αμφιβάλλω αν τα πράγματα ε, βελτιώθηκαν πολύ από το καθεστώ των ε, Ταλιμπάν και μετά, από την απελευθέρωση από το καθεστώ των Ταλιμπάν. Και ε, αυτή τη στιγμή ξέρω ότι υπάρχουν πάλι προβλήματα με του Ταλιμπάν και σχετικέ διαπραγματεύσει. Λοιπόν, απαιτούμε το δικαίωμα των γυναικών να τεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να ζητηθεί λογοδοσία, στο Αφγανιστάν από τις αρχές της χώρας αυτή, για τις διεθνεί του υποχρεώσει. Στο Πακιστάν, όπου είναι εύρωστη η κοινωνία των πολιτών, θα πρέπει να υπάρξουν γυναίκες ε, στις θέσεις εξουσίας. Είναι απαράδεκτο και ε, παράλογο να υπάρχουν απάνθρωποι, αντικοινωνικοί νόμοι κατά των γυναικών ε, για τους γάμους, την πλασφημία και το καθεξής. Θα πρέπει λοιπόν με το ψήφισμα αυτό να απαιτήσουμε λογοδοσία για την ε, κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό να καθορίζει τη σχέση και τη συμφωνία συνεργασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση με το Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Ευχαριστώ κύριε Γκόμε. Ο κύριο Σταβάρη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το Αφγανιστάν και το Πακιστάν είναι από τις περιπτώσεις που χαρακτηρίζουν τις χειρότερες τάσεις της ε, γεωπολιτικής ε, διεθνώς ε, και σε ταπικό επίπεδο. Βεβαίως υπάρχουν ακόμα χειρότερα προβλήματα. Εδώ λοιπόν οι χώρες αυτές προσωρινά είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή για τις διεθνείς πολιτικές. Υπάρχουν τάσεις φιλετικέ και αυτό είναι χαρακτηριστικό για το Αφγανιστάν, λόγου χάρη. Οι Ηνωμένε Πολιτείε εδώ και κάποια χρόνια βρίσκουν ότι δεν υπάρχει φιλετική λύση για το Αφγανιστάν. Εδώ και δεκαετίες, για να μην πω αιώνε και χιλιετίε είναι ιδιαίτερη κατάσταση τη χώρα αυτή. Εδώ λοιπόν ε, εξευρέθη η λύση, η τη μεταβατική κυβέρνηση με τη συμμετοχή των Ταλιμπάν, αλλά αυτό οδηγεί σε επιστοδρόμηση σε όλου του των κοινωνικών πρακτικών. Όπως η πώληση των γυναικών, ε, οι ομαδικοί βιασμοί για εγκλήματα τιμής κατά των οικογενειών, τέτοιες ε, πρακτικές κατά των γυναικών γενικότερα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε ότι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ευθύνη όταν εφαρμόζουμε τις συμφωνίες μα με τι χώρε αυτέ. Ευχαριστώ κύριε Ταβάρε. Ο συνάδελφος Ρέπο τελευταίο στη διαδικασία του Καρσία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κατάσταση των γυναικών στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν είναι άκρως ανισχυτική. Πριν από 10 χρόνια διεξήχθη η διάσκεψη του Πέτερσμπεργκ, όπου η διεθνής κοινότητα άρχισε να ε, οικοδομή ε, ελευθερίες, αλλά συνεχίζονται βιασμοί, αναγκαστικοί ε, γάμοι, βιοπραγίες κατά των γυναικών και ούτε η αστυνομία ούτε η δικαιοσύνη αντίδρα. Οι γυναίκες έχουν κατακτήσει κάποια θεμελιώδη δικαιώματα μεν, αλλά παραμένουν διακρίσεις σε ό,τι αφορά ε, την πρόσβαση στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό. Οι γυναίκες θα πρέπει να συμμετέχουν στην οικοδόμηση μιας δημοκρατικής και ανοιχτής κοινωνίας με ε, ενεργό τρόπο. Δεν μπορεί το Αφγανιστάν να αγνοεί το μισό του πληθυσμό. Η κατάσταση στο Πακιστάν ακόμα χειρότερη δυστυχώς. Ευχαριστώ κύριε Ρέπο. Για να ολοκληρώσει τη συζήτηση, το λόγο έχει ο Επίτροπος κ. Σαλμούνια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά το Αφγανιστάν, στη διάσκεψη της Βόνης πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τη διεθνή κοινότητα τόνισε και πάλι τη σημασία που αποδίδει στη διατήρηση των δικαιωμάτων των γυναικών η Πρόεδρος Άστον μαζί με την Υπουργό Εξωτερικών τον είπα, Χίρα Κρίντον συναντήθηκαν με Αφγανές στην αρχή της διάσκεψης ε, και πραγματικά μας εμπνέουν όλους μας οι γυναίκες αυτές. Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διαδικασία συμφιλίωσης θα πρέπει να ε, διατηρήσει και να επεκτείνει την πρόοδο που έχει κάνει η χώρα ήδη από το 2001 για τα δικαιώματα των γυναικών. Η κατάσταση των Αφγανών γυναικών στην κοινωνία αυτή συχνά παραμένει επισφαλής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το θέτει άμεσα υπόψη της κυβέρνησης του Αφγανιστάν όποτε έχει την ευκαιρία και τονίζει τη θέση της σε δημόσιες ε, δηλώσεις φέτος το Φεβρουάριο πούμε, για ξενώνε υποδοχή γυναικών στο Αφγανιστάν και πάλι το τόνισε στις ε, ε, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου τον Ιούλιο και τον ε, Νοέμβριο. Δικαιοσύνη και νομική συνδρομή για τις γυναίκες που πλήττονται από την ενδοοικογενειακή βία αυτό είναι έργο της Ένωσης. Ε, τα περαιτέρω θα εξαρτηθούν από τις ευρύτερες μεταρρυθμίσεις των θεσμών ε, του Αφγανιστάν. Συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και υποστηρίζει τις προσπάθειες στα της διαδικασίας λεγόμενης Καμπούλ. Για το Πακιστάν τώρα. Η πρόθεση των δικαιωμάτων των ε, γυναικών είναι προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη έχουν δεσμευτεί στην κατεύθυνση αυτή με το Πακιστάν. Η πρόοδος θα εξαρτηθεί από τη δράση της κυβέρνησης της χώρας αυτής, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη μπορούν να ασκήσουν πίεση ε, με το διάλογο, με την κυβέρνηση, υποστηρίζοντας μέτρα ε, και βοηθώντας γυναίκες για την πρόσφυγή τους στη δικαιοσύνη πολλά προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν οι γυναίκες. Μεταξύ αυτών είναι η βία ε, το σοβαρότερο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συστηματικά χρησιμοποιεί τον πολιτικό διάλογο με το Πακιστάν για να ε, φέρει στο επίκεντρο τέτοια ζητήματα για την ενεργή υλοποίηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για άρση των διακρίσεων κατά των γυναικών που έχει υπογράψει και το Πακιστάν και είναι ενεχόμενο μέρος. Θα πρέπει να εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία, να καταστεί παράνομη κάθε είδους βία κατά των γυναικών και να υποστηρίζονται τα θύματα της βίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Αλμούνια. Έχουν κατατεθεί συνολικά 7 προτάσεις ψηφίσματος όλων των πολιτικών ομάδων. Ολοκληρώνεται η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει μετά το τέλος της επόμενης συζήτησης ε, που ακολουθεί τώρα και είναι για